Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και για το έργο που επιτελέσατε εδώ σαν αυτό το θέμα. Ευχαριστώ συνάδελφο και τώρα εδώ κλείνει η παρούσα συζήτηση. Λέει ο πρόεδρο και τώρα προχωρούμε ή στο επόμενο θέμα τη μέσα διάθεση που είναι η σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση με συντάκτη των Κάρλ Χάιντ Φλόρεν για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο εισηγητή το λόγο, αρκεί να βρίσκεται στην αίθουσα. Καλ Χάιντ, απ, εκεί είσαι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ξεκινήσω κοινότοπα, να πω στους συναδέλφους ε, ε, τι εννοούμε όταν μιλάμε για ηλεκτρικά απορρίμματα, γιατί όλοι μας λένε, πολλοί μας λένε ότι είναι επουσιώδη αυτά. Ένας τόνος ηλεκτρικών απορριμμάτων ε, περιέχει ένα εκατο... Συγγνώμη, ένα εκατομμύριο ε, κινητά τηλέφωνα έχουν 24 κιλά ε, παλάδιο, χρυσό, 9 τόνους ε, χαλκό, ένα τόνο. Ένας τόνος κινητά, κύριε Πρόεδρε, έχει 50 πιο, φορές πιο πολύ χρυσό από ότι ένας τόνος γης. Γι' αυτό λοιπόν καθίσταται σαφές πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για τις πρώτες ύλες και πόσο εύκολα ε, εξάγουμε και διώχνουμε τέτοια απορρίμματα από την Ευρώπη στην Αφρική όπου τη χάνει μεταχείριση με καταστροφικό τρόπο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τις τιμές αυτές και γι' αυτό χάρηκα που συμφωνήσαμε σε βασικές ε, αρχές στην οδηγία αυτή, οι οποίες πήραν το σωστό δρόμο. Η παράνομη ε, διοχέτευση των υλικών αυτών ε, είναι σημαντικό θέμα. Έχουμε το ερώτημα όμως κατά πόσον τα κράτη-μέλη είναι πραγματικά σε θέση και διτεθειμένα και αυτό ισχύει και η δική μου χώρα να πράξουν τα απαραίτητα, να διαθέσουν το απαραίτητο προσωπικό προκειμένου ο κανονισμός αυτός να περάσει και να εφαρμοστεί και στα τελωνία και στους λιμένες. Ένα άλλο βασικό ζήτημα που πετύχαμε είναι οι στόχοι για την συλλογή που είναι σημαντική. Στην Σουηδία 16 κιλά και σε μία νότια χώρα από που προέρχεται το όνομά μου 30 κιλά. Είναι μεγάλη καταστροφή αυτή σε, πολλούς, σε πολλές ε, ιδρύτριες χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ε, ποσά 3-4 κιλά κατά κεφαλή. Πρόκειται για ντροπιαστικά, για ντροπιαστικούς ρυθμούς. Όλους αυτούς τους στόχους συλλογή τους πετύχαμε ευτυχώς. Δυστυχώς το Συμβούλιο είναι πολύ φλεγματικό το έργο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ξαναείδαμε αυτό σε όλες τις διαπραγματεύσεις δεν αποδειχθηκε διτραφυλικό προς την Ευρώπη. Αν παράγεται ένας λαμπτήρας από μία επιχείρηση στην Ευρώπη, θα πρέπει κάποια στιγμή να περάσει στην ανακύκλωση. Θα πρέπει να κάνει κανείς ε, ως επιχειρηματίας ε, αίτηση σε 27 διαφορετικές χώρες με διαφορετικά συστήματα για την ανακύκλωση. Για τον ε, ΦΠΑ μπορεί να κάνει κανείς μία αίτηση. Όχι όμως. Για τους λαμπτήρες επιβαρύνονται έτσι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ένα λαμπτήρα. Αυτό από μόνο του κοστίζει 60 εκατομμύρια ευρώ αναχρόνω για κάθε διαδικασία. Μειώσαμε κάπως τη γραφειοκρατία, εν πάση αλλά το Συμβούλιο στα θέματα αυτά μένει σε αυτά τα μεγάλα ποσά που πληρώνουν οι επιχειρήσεις και το Συμβούλιο φυσικά δεν θέλει να αγγίξει τα τεράστια αυτά χρηματικά ποσά. Κι όμως αυτά μπορούν να διοργανωθούν με πολύ πιο εύκολο τρόπο τεχνολογικός πώς. Κύριε Ποτότσνικ, λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να σας είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη διαδικασία αυτή διαδραματίσατε πολύ σημαντικό ρόλο. Αν δεν ήσασταν εκεί, θα είχαν αποτύχει οι διαπραγματεύσει αυτές. Το Συμβούλιο τοποθετήθηκε με τρόπο που δεν έχω ξαναγνωρίσει τα 22 αυτά χρόνια και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να εξαρέσω τη χώρα μου. Η βούληση σύνδεση της ε, οικολογικής ε, πολιτικής με οικονομικά κριτήρια χρησιμοποιείται για εσωτερική πολιτική. Ούτε καν τον ορισμό της ανακύκλωσης μπορέσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να τον ορίσουμε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Η κατεύθυνση είναι σωστή, αλλά πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν για να στραφούμε προς την κατεύθυνση και εννοώ πολλούς, όχι μόνο ένα-δύο κρατημέλη. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κ. Ποτότσνικ, εκ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μικροφόνο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Έχουμε δύο σημαντικά ζητήματα στην ατζέντα σήμερα. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερω τον εισηγητή και τον κύριο Καλ Χάιντ Φλόρεντς και τους Κιώδη. και τις ομάδες τους για την επιτυχία στι διαπραγματεύσει για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στάθηκαν το ένα δίπλα στο άλλο στη συζήτηση αυτή για να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι, για να μειωθεί σαφώς το διοικητικό άκτος και να δοθούν αρμοδιότητες ε, στις ε, αρχές των ευρωπαϊκών ε, κρατών σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές. Ως τώρα πετύχαμε και χαίρομαι γιατί η προτινόμενη οδηγία πετυχαίνει σε μεγάλο βαθμό τους στόχους που είχε ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που ήθελε να πετύχει με την πρόταση που κάναμε. Ασφαλώς θα ήθελα να κινηθούμε πιο γρήγορα και να κινηθούμε και περαιτέρω, όπως ανέφερε και ο κύριος Φλόρεντς. Και είμαι βέβαιος ότι το ίδιο επιθυμείτε και πολλοί από εσάς. Αλλά σαφώς δίδεται μια νέα ορμή, μια νέα, μια νέα δυναμική σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό και το ηλεκτρικό απορρίμματα και θα πρέπει να την υποστηρίξουμε. Να σας δώσω μία ιδέα για το τι επίπεδο βελτίωση ε, θα πετύχει η, τρέχουσα, η οδηγία αυτή σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση. Ένα γρήγορο υπολογισμό. Ο στόχος συλλογής είναι 4 κιλά κατά κεφαλή κατά έτος κατά κράτος μέλος με 500.000 500 εκατομμύρια κατοίκους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι 2 εκατομμύρια 2 ε, εκατομμύρια τόνους ε, από τα 10 εκατομμύρια τόνους ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απορρίμματα πρέπει να συλλέγουν τα κρατημέλη. 20%. Η νέα οδηγία θα υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να συλλέγουν το 85% των απορριμμάτων αυτό. Άρα μέχρι το 2020 υπολογίζουμε ότι θα είναι 12 εκατομμύρια τόνοι που θα απορρίπτονται το χρόνο. Θα πρέπει να συλλέγουμε 10 εκατομμύρια εξ αυτών μέχρι το 2020. Μόλιβδος, χρώμιο, κάδμιο, υδράργυρο, τα οποία θα τη χάνουν σωστής επεξεργασίας. Ε, χρυσός, ε, πλατίνιο, χαλκός. Όλα αυτά θα πρέπει να διοχετεύονται και πάλι στην ε, αλυσίδα παραγωγής και να μειώνονται έτσι το κόστος παραγωγής και οι εκπομπές. Μπορεί να μην είναι πολύ επιστημονική αυτή η υπολογισμή, αλλά μας καταδεικνύουν ότι κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός με την, τρέχουσα, με την οδηγία αυτή. Χρειάζεται η σωστή επεξεργασία των υλικών αυτών προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Μας ανησυχούν ιδιαίτερα μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε τρίτες χώρες, επιζήμιες για το περιβάλλον και τον ανθρώπινο οργανισμό. Κατά το παρελθόν υπήρχαν διάφορες ε, τέτοιες καταχρήσεις ε, σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές απορριμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται στα διεθνή φόρα για να αποτρέψει νόμιμες οδούς για την ε, αποστολή χρησιμοποιημένων υλικών. Να σας πω σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποδέχεται το κείμενο το οποίο διαπραγματεύτηκαν ε, τα θεσμικά όργανα και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να διασφαλίσει την πλήρη και ομαλή εφαρμογή μετά την έγκριση από πλευρά του Κοινοβουλίου και από πλευρά τη Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε κάποιε δηλώσει για να συνοδεύσει αυτές τις, ε, την έγκριση. Καταρχά, ε, ό,τι αφορά το σχεδιασμό των προϊόντων, σε ό,τι αφορά τις σχετικές προϋποθέσεις σύμφωνα με την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού. Κατά δεύτερον, μεταβατικές ε, ρυθμίσεις για τα κράτη-μέλη θα πρέπει να περιοριστούν σε εξαιρετικές ε, ε, περιπτώσεις για τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να είναι αντικειμενική η αξιολόγηση και να υπάρχει δυνατότητα απόδειξης τους Τρίτον, τα νανοηλικά θα πρέπει να υπάγονται στη γνωρισμό των νανοηλικών που περιλαμβάνεται στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενδεχόμενοι κίνδυνοι θα πρέπει να ορίζονται και από τη σχετική νομοθεσία. Τέταρτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι προκειμένου να υπάρχει συνοχή με τη συνθήκη, οι αρμοδιότητες που έχει για την ε, μεθοδολογία υπολογισμού σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και σε ό,τι αφορά την ε, καθιέρωση επιπλέον ε, κανόνων θα πρέπει να γίνεται με καταξιοδότηση πράξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο ότι επιφυλάσσεται της δυνατότητας να λάβει τα σχετικά μέτρα και να ζητήσει δικαίωση από το ΔΕΚ. Και τέλος, Πρέπει να σας πω κυρίε και κύριοι, αγαπητοί βουλευτές, ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικές ε, και ηλεκτρικές συσκευές αποτελούν έναν αυξανόμενο όγκο που περιλαμβάνει σπάνια μέταλλα, σπάνιες ύλες που αξίζουν να ανακυκλωθούν. Τα απορρίμματα αποτελούν πραγματικά έναν πόρο. Αυτό κατήσατε όλο ένα και πιο σοφές και θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Σωστά ακούσατε, δεν πρόκειται μόνο για θέμα περιβαλλοντικής συντήρησης, πρόκειται για ένα από τα βασικά ζητήματα για την ανταγωνιστικότητα της ε, μελλοντική ευρωπαϊκής οικονομίας. Σας ευχαριστώ. Zebra, have the floor. Ο κύριος Σέμπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καρλ Χάινς ε, Φλόρενς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά που κάναν. Πρόκειται για μια αναδιατύπωση και όπως ξέρουμε η υφιστάμενη οδηγία στις 13 ε, ε, τέθηκε σε εφαρμογή το 2013, πριν από 10 χρόνια σχεδόν και λίγα πέτυχε ουσιαστικά ο Καρλ Χάινς μας ανέφερε πόσο μεγάλες διαφορές υπάρχουν μεταξύ των ε, κρατών μελών. Στη Ρουμανία 0,8% κιλά, 7,8 κιλά κατά κεφαλή στη Γερμανία. Είναι πάρα πολύ μεγάλες διαφορές και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν καταφέρουμε στην οικονομία μας ε, να δημιουργήσουμε μια τέτοια κυκλοφορία δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν επαρκεί ε, πόροι σε ό,τι αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό, όπως είπε ο επίτροπο, η αξιοποίηση μετά τη χρήση του προϊόντος θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη φάση του σχεδιασμού. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Αυτή η οδηγία είχε κάποιε αδυναμίες. Ε, έλειπε, για παράδειγμα, αυτό ο σύνδεσμό με τον οικολογικό σχεδιασμό η σημερινή ε, οι σημερινοί στόχοι που τύφονται με την ε, νέα οδηγία για το 85% είναι σαφώς πιο σωστή. Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθούν αποτελεσματικά συστήματα συλλογής και αυτό εξαρτάται και από τα κράτη-μέλη προκειμένου να δώσουν μια χείρα βοηθείας προς τον καταναλωτή προκειμένου ο καταναλωτής να έχει δυνατότητα να κάνει κάτι από μόνος του. Νομίζω ότι συνολικά θα εξαρτηθεί και από τα κράτη-μέλη πώς θα εφαρμοστούν τα συστήματα. Έχω εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρόκειται να τα παρακολουθήσει όλα επακριβώ προκειμένου να πετύχουμε του συνολικού στόχου, γιατί σε μακροπρόθεσμο επίπεδο είναι η μοναδική ευκαιρία που έχουμε για να διατηρήσουμε το περιβάλλον μα. Ευχαριστώ κυρία Φαμπρέντ. Ευχαριστώ πρόεδρε συνάδελφοι. Κάποιος είχε πει στο τέλη του 19ου αιώνα αν θέλεις να γίνεις πλούσιος θα πρέπει να κατασκευάζεις σε προϊόντα τα οποία ο κόσμος τα πετάει μετά τη χρήση και νομίζω ότι τότε δεν αντιλήφθηκε ότι ξεκίνησε μια κουλτούρα του πετάγματος. Αυτό αποτελεί σύμβολο και μεγάλο πρόβλημα σήμερα. Και όταν το 2003 τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά η οδηγία, εστιαστήκαμε στα προβλήματα της ε, κοινωνίας αυτής της μία χρήσης το θέμα της ποιότητας του εδάφους, της ατμόσφαιρας, η κοινωνικός αντίκτυπος ε, της κακής ανακύκλωσης ε, στα Στι χώρε του τρίτου κόσμου και επαναλαμβάνω ότι αυτά τα επιχειρήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά αλλά όπως είπε και ο Επίτροπος μάλλον θέλω να προσθέσω ένα επιχείρημα σε ό,τι αφορά τα ευγενή μέταλλα τα οποία βρίσκονται στα κινητά μα τηλέφωνα και σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μας υποστήριξε και η ίδια η βιομηχανία στην αναθεώρηση αυτή, στην αναδιατύπωση αυτή υποστήριξη την οποία λάβαμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία όμως δεν λάβαμε δυστυχώς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι κανόνες σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μόνο καλοί, αλλά και απολύτως απαραίτητοι. Θέλουμε υψηλούς στόχους για την ανακύκλωση, θέλουμε να φροντίσουμε τα μικρές συσκευές ε, που περιέχουν πολύ σημαντικά υλικά να υπάρχονται σε υψηλούς στόχους. Τέλος. Θα ήθελα και αυτό το λέω με απόλυτη υπεποίθηση να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον εισηγητή που κατάφερε να προωθήσει την θέση του Κοινοβουλίου με ένα συμβούλιο το οποίο όπως σας είπα κυμαίνεται σε λάθος μήκος κύματος και είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι θα υπερψηφιστεί αυτό το αποτέλεσμα από την ομάδα μου αύριο. Thank you, Κύριε Παναγιώτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Συνάδελφοι. Αυτή η συμφωνία επί της νέας οδηγίας είναι το αποτέλεσμα μακρών και δυσκόλων διαπραγματεύσεων. Και με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο, τον κύριο Πότουτσνικ, για την κατανόηση, για το πώς αφοσιώθηκε σε το θέμα, αλλά και τον Καρλ Χάιτς Φλόρενς, τον εισηγητή, για την αφοσιωτικότητα που έδειξε επίσης, για να πετύχουμε το τελικό θεωρητικό, θετικό αποτέλεσμα, γιατί έτσι νομίζω ότι έχουμε θέσει τα θεμέλια, ούτως ώστε ε, να, να μπορέσουμε να έχουμε σωστή διαχείριση αυτών των αποβλήτων. Περίπου 30% τώρα έχουμε ανακύκλωση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται. Γιατί το 30% ανακυκλώνεται, το 70% μένει ή στις χωματερές ή παρανόμως ε, ε, διοχετεύεται Με τη νέα οδηγία όμως έχουμε τις απέτες συνθήκες ώστε να έχουμε μία και, νέα και κοινή αγορά για αυτά τα απόβλητα. Έξι χρόνια από τότε που ξεκίνησε η υπόθεση, δηλαδή το 2018, όλα αυτά τα απορρίμματα θα έχουν καλυφθεί. Και έχουμε και άλλους στόχους ακόμα πιο φιλοδόξους. Με το 2019 θα πρέπει 65% να περισυλλέγουμε από όλα αυτά τα απόβλητα Όλα αυτά τα οποία κατελήγουν στην αγορά τώρα και κάποια άλλη ε, καινοτομία είναι το ότι προσπαθούμε να δούμε πώς ε, θα έχουμε πιο αποτελεσματικές ε, συνθήκε και πολιτικές ούτως ώστε να δούμε πώς θα έχουμε 400 τετραγωνικά ούτως ώστε να μπαίνουν πώς ανακύκλωση αυτά τα υλικά. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά υπέρ η οδηγία. Είναι κάτι που όλοι μαζί το πετύχαμε και είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει όλους και θα ωφελήσει και κυρίως για το μέλλον. Ο Στρεμόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριοι συνάδελφοι είμαστε ένα βήμα πριν από μια σημαντική συμφωνία για τη βελτίωση της διαχείρισης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. μετά από μια ενδελεχή διαδικασία διαβούλευσης με την επιτροπή και το συμβούλιο καταλήξαμε σε ένα κείμενο συμβιβαστικό το οποίο εμείς στηρίζουμε ως πράσινοι. δεν είναι μια ριζική αντιμετώπιση του ζητήματος αλλά σίγουρα είναι ένα σημαντικό βήμα σαν ε, ομάδα των πράσινων πιέσαμε ιδιαίτερα να αυξηθούν οι στόχοι συλλογή και να υπολογιστούν στη βάση των αποβλήτων που προκύπτουν να υποχρεωθούν οι διανομείς να συλλέγουν τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα χωρίς καμιά υποχρέωση αγοράς από τον καταναλωτή καθώς και για αυστηρότερους ελέγχους των ε, αποβλήτων αυτών σε ό,τι αφορά την επαναχρησιμοποίησή τους και την εξαγωγή τους σε χώρες εκτός οσα ήμασταν η μόνη ομάδα που έκανε προτάσει σχετικά με τα νανοηλικά. δεν καταφέραμε να αποσπάσουμε την δέσμευση των παραγωγών να αναφέρουν την ύπαρξη των νανοηλικών πάνω στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα αλλά καταφέραμε να πείσουμε την επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσο είναι απαραίτητη η επιλεκτική επεξεργασία των νανοηλικών στα απόβλητα αυτά. εύχομαι το κοινοβούλιο να ψηφίσει θετικά και βέβαια να αντιμετωπίσει τη χαμηλή ε, συλλογή τα χαμηλά ποσοστά τη βελτίωση της διαχείρισης και της επεξεργασίας καθώς και τον έλεγχο των παράνομων εξαγωγών των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων σε τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ χαίρομαι που αναλάβατε ξανά την διάθεση των συζητήσεων και θα ήθελα να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου ε, ε, αυτή η αναβάπτιση του νομοθετήματος ε, είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας των κρατών μελών να μπορέσουν να συγκροτήσουν κάποια συστήματα ανακύκλωσης για αυτά τα υλικά 2003-2008 προβλεπόταν. Κοιτάξτε, το 2008 είχαμε πει ότι 70% των ηλεκτρονικών ε, τα οποία αντί να γίνεται τίποτα άλλο πάλι εξήγουν το παρανόμος ή μένανε ή στις ε, χωματερές και όλοι συμφωνήσαμε ότι αυτό είναι τραγικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να δούμε οι πράσινοι τι κάνανε. Πάντως νομίζω ότι ο Καλ Χάιντς Φλόρεντς ε, δούλεψε πάρα πολύ σκληρά και έτσι απέσπασε αυτή την πάρα πολύ ευμενή λύση. Τώρα έχουμε κάποιες μεταβολές, τις χαιρετίζουμε και θεωρούμε ότι θα βοηθήσουν τόσο να βελτιθεί η κατάσταση οι σχετικοί στόχοι έχουν προσαρμοστεί ε, και όσο, όσον αφορά τη μεθοδολογία και όσον αφορά το ύψος του, του, του πύχη ε, κάποια κρατημέλη έχουν θέσει άλλο timing αλλά ε, αυτό που χρειάζεται περισσότερο χρόνο θα κάνει πιο αποτελεσματικό και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη ότι τα κράτη-μέλη μπόρεσαν να κάνουν ρυθμίσει αυτόνομε, ιδίω για τη χρηματοδότηση και έτσι να αποφύγουμε κάποιο είδου ε, αύξηση του κόστους για τις κοινωτικές και δημοτικές αρχές όμως τώρα έχουμε το θέμα της ε, υπευθυνότητας γιατί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα της ανακύκλωσης οι ιδιώτες. Ιδίω όπως έχουμε σήμερα το πρώτο μας θα πρέπει να έχουμε τις ε, παρέντες πληροφορίε για τα κρατημέλη τώρα έχουν ένα το πλαίσιο τους ώστε να αποδώσουν καρπούς οι προσπαθειές τους τώρα τον μπαλάκι στο γήπεδο τους για να κάνουν αυτή πετύχουν κάποιο αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστώ και εγώ για τα καλά σα λόγια. Πάρα πολύ χαίρομαι που οι γυναίκε χωριέ ομάδα είναι με το μέρο μου και ο επόμενο παραγωγητή είναι η κυρία Βίλ. Εδώ και καιρό συζητάνε τέτοια ζητήματα τα αναπτυσσόμενα, τα αναπτυγμένα κράτη. Θα σας προκαλέσει έκπληξη ότι ζούμε όπως ζούμε εις βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών βασική, βασικό θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, ανοιχτός τομέας εφαρμογής. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για την νομοθεσία. Χαίρομαι που τέθηκε ο στόχος του 85% για όλους, γιατί το Συμβούλιο προσπαθούσε να πετύχει χαμηλότερους στόχους και πολύ επίμονα. Το Κοινοβούλιο, το λέω πάντα, θα πρέπει να ασκεί πίεση, γιατί αν ασκείται τέτοια πίεση θα γίνονται και ανάλογες επενδύσεις. Και χαιρετίζω στο πλαίσιο αυτό το γεγονός ότι τα ηλιακά στοιχεία δεν αφαιρέθηκαν από την οδηγία. Καλό ήταν που δεν ε, μείναμε στο επίπεδο εθελούσιας δέσμευσης των παραγωγών, γιατί στο παρελθόν είχε υποκύψει σε πιέσεις τέτοιες ανάλογες στο Κοινοβούλιο. Και σε τελική ανάλυση αποτελούν μόνο ένα εργαλείο της καθυστέρησης. Δεν συμφωνώ, ωστόσο, για το πώς αντιμετωπίζονται τα νανοηλικά στην οδηγία. Θα πρέπει οι παλιές συσκευέ με νανοηλικά να τη χάνουν διαφορετικής μεταχείρισης. Ωστόσο, στην έκθεση καλείται απλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον αυτό θα πρέπει να συμβεί στο μέλλον. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί εξαιρετικά ήπια διατύπωση που δεν αξίζει τίποτε τα νανοηλικά θα, μπορούσαν να είναι, θα μπορούν να είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον και για, και για τον άνθρωπο, για την υγεία του ανθρώπου. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει ε, επακριβώς τα νανοηλικά σε περίπτωση που δεν αποδειχτεί ότι είναι αυλαβή για τον οργανισμό, δεν θα πρέπει να τους δοθεί άδεια να κυκλοφορούν στην αγορά η αιμονή του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις απέδωσε καρπούς ωστόσο και θα ήθελα γι' αυτό να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η οδηγία επιβάλλει την επιλεκτική ανακομιδή των ηλεκτρονικών συσκευών και κατά συνέπεια την ανακύκλωση. και υπάρχει το κόστος εις βάρος των παραγωγών, ε, υπάρχει υποχρεωτικό ποσοστό 5% για την, για την επαναχρησιμοποίηση και προβλέπει όμως ε, για τις μικροσυσκευές την ανακομιδή ε, στους μικρούς, στην έδρα των μικρών παραγωγών. Το σύστημα αυτό δε ίσχυε όμως και για τα μικρά μαγαζιά. Για να μπορεί να έχουμε όμως ένα τέτοιο σύστημα περί δεν θα πρέπει τα κράτη-μέλη να επιτρέπουν μη αναγνωρισμένους χρήστες να παίρνουν τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές σύσκευες, οι οποίες βγαίνουν έτσι από το κύκλωμα. Η κυρία Γκαρντίνη, μιλάμε σίγουρα για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, όπως ε, θύμισε ο κύριος Φλόρενς, ε, μιλάμε για επικίνδυνα ρηπογόνα προϊόντα για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία. Μιλάμε όμως και για μια καταπληκτική δυνατότητα ε, ανασυλλογής πολυτίμων ουσιών και έχω κατά νου το ίμβιο το οποίο στοιχίζει χιλιάδες επί χιλιάδων ευρώ το, γραμμάριο. Τώρα αναφερόμενοι στη χώρα μου πράγματι δεν έχει τα επίπεδα της Βορείου Ευρώπης όπου η ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών είναι πολύ σημαντική αλλά όμως έχουν γίνει σημαντικά βήματα με βέβαια ανομοιογένειες ε, στην ε, επικράτεια στο βορρά έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό η περιοχή μου το, ε, το Βένετο έχει ξεπεράσει τα όρια είναι στην τρίτη θέση με τον Μπελούνο πάνω από όλους και η Εμίλια Ρωμάνια είναι 100%. Ε, πρόκειται για πλήρη κάλυψη. Η τάση είναι πολύ σημαντική. Τα τελευταία χρόνια είχαμε αύξηση 27%. Θα πρέπει να κρίνουμε θετικά το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, ο δρόμος που έχουμε πάρει είναι ο σωστός, πρέπει να προχωρήσουμε σε μία ε, καμπάνια πληροφόρησης ε, προς τους πολίτες και να ενισχύσουμε όλες εκείνες τις διαρθρώσεις οι οποίες είναι ήδη ενεργές και να ενημερώσουμε και τα στοιχεία εκείνα τα οποία, δεν, ε, τα οποία μας εμποδίζουν να έχουμε γρήγορη εξέλιξη. Η κυρία Σάρμπου.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 είναι πηγή προβλημάτων. Ε, είναι κάτι το οποίο έχει φουσκώσει, έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια γιατί πρόκειται για πάρα πολύ επικίνδυνα απόβλητα και απορρίμματα αυτού του είδου. Διότι δεν, δεν, δεν, δεν την χάνουν ορθή διαχειρήσεω και καταλήγουν στι χωματερέ και αποτελούν ουσιαστικά τοξικά απόβλητα. Έχουμε εδώ την ε, σχετική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ώστε ε, να υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση. Αυτό είναι κάτι οποίο το χαιρετίζουμε. Όμω η κατάσταση διαφέρει από χώρα ει χώρα. Οπότε θα πρέπει αυτή η πραγματικότητα να ληφθεί υπόψη και έτσι η νομοθεσία να καταστεί αποτελεσματική και να είναι ευκόλως εφαρμόσιμη. Διότι ή στην Ρουμανία η αγορά των ηλεκτρονικών προϊόντων δεν έχει ακόμη κοριστεί. Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τόσο πολλά ε, τέτοιου είδου απόβλητα όπω Οπότε για μα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε περισσότερο χρόνο τόσο ώστε να μπορούμε να προσαρμοστούμε ει αυτού του ε, φιλοδόξου ή στόχου οι οποίοι έχουν τεθεί. Και όσον αφορά την ανακομιδή. Ε, έχουμε κάποια βελτίωση τα τελευταία 7 χρόνια και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και ταυτοχρόνως ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα ε, έχουμε κάποια ισορροπία μεταξύ στόχων και πραγματικότητα. Εγώ πάντως θα πρέπει να ευχαριστήσω εισηγητή και σκιώδης εισηγητάς για την δράση την οποία ανέπτυξαν κατά τις τόσο δύσκολες διαμονές με το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον, ε, και να συγχαρώ τον Καρλ Φλόρεντς γιατί για την το έργο του. Πάνω από τρία χρόνια αυτός και η Επιτροπή του εργαστήκαν για το θέμα αυτό. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που πολλοί συναδελφοί ανέφεραν, αλλά θα ήθελα να τονίσω ένα μικρό ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες ωστόσο, γιατί σε ενεργειακούς φλαμπτήρες οι οποίοι ε, εξοικονομούν 80% του ηλεκτρισμού σε σχέση με τους άλλους λαμπτήρες, αλλά περιλαμβάνουν σπάνιες γιές, τις οποίες θα πρέπει να τις ανακτούμε και είναι... περιλαμβάνουν πολύ... περιλαμβάνουν υδράγυρο. Πολύ λιγότερο από ότι τα θερμόμετρα που χρησιμοποιήσαμε μέχρι πριν από κάποια χρόνια, αλλά θα πρέπει να απορρίπτεται και να κυκλώνεται με σωστό τρόπο. Στην ε, πόλη μου ήθελα να απορρίψω μικρές συσκευές και μου είπαν να τα βγάλω εκτός πόλεως ε, τη Δευτέρα ε, μέχρι τις 3.30. Ε, είμαστε μόνο ανοιχτά. Μα ποιο άνθρωπο που δουλεύει έχει χρόνο την Τρίτη μέχρι τις 3.30. Γι' αυτό λοιπόν υποβάλαμε ένα αίτημα προκειμένου να υποχρεωθεί το κατάστημα να λαμβάνει τις χρησιμοποιημένες σε αυτές τις συσκευές και τους λαμπτήρες. Χάρηκα που πέρασε αυτό και το πέρασε ο Καλχάιτ Φλόρεντς. Είναι μια ένδειξη ότι λαμβάνουμε στα σοβαρά τους πολίτες και ότι τους διευκολύνουμε την επιστροφή τέτοιων συσκευών προκειμένου να την χάνουν σωστής ε, αντιμετώπισης. Ευχαριστώ πολύ και τώρα η κυρία Μερκής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή ο οποίος ε, τα κατάφερε εξαιρετικά γιατί το έργο του δεν ήταν και εύκολο. Πετάμε τα ευγενή μέταλλα. Και σε τέτοιες εποχές κρίσης δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το πράττουμε αυτό. Σύγχρονες συσκευές ε, όπως τα κινητά τηλέφωνα βρίσκουν από τέτοιες από τέτοια υλικά τα οποία τα χρειαζόμαστε. Το θέμα είναι η συλλογή, αλλά όχι μόνο η συλλογή. Γιατί αν ένας χασάπης, για παράδειγμα, ανοίξει ένα κινητό, δεν πρόκειται να έχει τα αποτελέσματα που θα έχει ένας ειδικό. Θα πρέπει λοιπόν να αφαιρούμε αυτά που θέλουμε να αφαιρέσουμε και γι' αυτό λοιπόν στην συλλογή θα πρέπει να κοιτάξουμε πολλές πτυχές της διαδικασία. Θα πρέπει να κοιτάξουμε ποια είναι τα καλύτερα και πιο ποιοτικά αποτελέσματα και όχι τον πιο εύκολο δρόμο. Να τα πετάμε δηλαδή σε άλλε χώρε, το οποίο είναι επιβλαβέ για το περιβάλλον και δεν μα αποφέρει αυτά που θέλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Βίμπνερ. Κυρία Βίμπνερ, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Καρλ Χάιντ Φλόρεντ επετέλεσε έργο πάρα πολύ σημαντικό. Όλα όσα έκανε σε σχέση με αυτή την έκθεση απίτησαν πάρα πολύ προσεκτική εργασία. Συνήντησε πολύ κόσμο, μίλησε με πάρα πολλούς. Δυστυχώς βέβαια υπήρξαν ε, αποκλίνω στις απόψεις. Πάντως, ο στόχο ήταν κοινό. Δηλαδή το πώ θα μειώσουμε τον όγκο αυτών των ε, απορριμμάτων και αποβλήτων. Αυτά τα οποία έχει αντιμετωπίσει τώρα η Ευρώπη. Οπότε, με το έγγραφο αυτό κάνουμε κάτι σημαντικό. Ε, γιατί λέμε πώ είναι δυνατόν να έχουμε εξοικονόμηση πόρων. Και ταυτοχρόνω, αυτό το οποίο κάνουμε είναι τη, να, να αξιοποιήσουμε αυτά τα απόβλητα. Επίσης, εδώ στην Ευρώπη έχουν πάρα πολλές δυσκολίες όσον αφορά τα... Ε, ε, τις πρώτες ύλες. Να, επομένως εδώ πέρα κάποιες ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε. Οι πρώτες ύλες μπορούν να προέλθουν από αυτά τα απορρίμματα, αυτά τα απόβλητα. Άρα να μην πηγαίνουν αυτά τα είδη ή στην χωματερή. Επίσης, μπορούμε να παρατείνουμε την ζωή, την περίοδο χρήσεως των, των ε, προϊόντων. Πολλές φορές γίνεται ανταλλαγή του παλαιού με το καινούργιο. Οι προβλημόνες κυρώσεις είναι το τελευταίο καταφύγιο. Το πιο σωστό είναι πρώτα να χρησιμοποιήσουμε τις άρεστες πρακτικές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για πολύ καιρό παρήγαγαν οι Ευρωπαίοι απόβλητα χωρίς να ανησυχούν για την ανακύκλωσή τους. Σήμερα ακόμη οι ελάχιστοι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την, ε, την αντίδραση, έχουν το ρεφλέξ ε, για να ανακυκλώνουν ε, τις ηλεκτρικές τους συσκευές. Εγώ το περασμένο Σαββατοκύριακο θέλησα να δώσω για ανακύκλωση ένα πολύμπριζο στο μαγαζί, σε ένα μαγαζί. Και δεν ήξερε ο υπάλληλος τι να κάνει. Ο υπεύθυνο του εξήγησε ότι υπήρχε ε, ένας κάδος ειδικό για την ανακύκλωση μέσα στο μαγαζί. Δεν το ήξερε ο υπάλληλος. Μόνο το 33% των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων ε, μαζεύεται σήμερα ε, και ανακυκλώνεται. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Καρλ Χάιτς Φλόρεντς για τη δουλειά του και τον ευχαριστώ γιατί ορίζει το στόχο για κάθε κράτος μέλος ένα ποσοστό περισυλλογής ε, μέχρι το 2013 ε, στην κάθε, χώρα ε, και δίνει την δυνατότητα διότι οι κάδοι περισυλλογής αυξάνονται και υπάρχει και μία ε, βαθμιαία προσέγγιση της στην περισυλλογή των προϊόντων προς ανακύκλωση. Αγαπητοί Ευρωπαίοι πολίτες, ας διαλέγουμε τα σκουπίδια. Αυτό είναι καλό για μας και για τις επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ. Και σας παρακαλώ επίσης να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να κατεβάσουμε τη θερμοκρασία του κλιματισμού διότι σε αυτό το ημικύκλιο κάνει κρύο και σπαταλούμε και ενέργεια. Ευχαριστούμε και τόσο υποτελεί ο Πρόεδρος. Έχετε το λόγο. Δεν το κάτσετε. Πρώτα ευχαριστώ, συγχαρητήρια στον Καρλ Χάιντ. Είναι συνάδελφος και δεν είναι μέλο των Πρασίνων, από ό,τι βλέπω και το ΕΛΚ επιτελεί σημαντικό έργο για τα θέματα αυτά. Τώρα, ε, όσον αφορά αυτά τα απο, απορρίμματα, τα απόβλητα, ε, έχουμε εδώ πέρα σημαντικό κίνδυνο για την δημοσία υγεία. Και ε, ο όγκος τέτοιων απορριμμάτων αυξάνει συνεχώς. Θα πρέπει επομένω με αίσθημα ευθύνη να θεσπίσουμε την αποτυμένη νομοθεσία που να οδηγεί στην ανακύκλωση. Άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κρατημέλη να μπορέσουν να καθοδηγήσουν τι επιχειρήσει για το τι θα κάνουν για να έχουμε καλύτερη διαχείριση των σχετικών πόρων. Οπότε να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε με την ανάκτηση του σχετικού υλικού όλων αυτών των ε, μηχανημάτων. Να δούμε πώ θα έχουμε αηφόρο παραγωγή, πώ θα έχουμε ευθύ ανάκτηση και ανακομιδή αυτών των απορριμμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt deșeurile cu potențialul cel Ευχαριστώ πολύ. Τα απορρίμματα αυτά αυξάνονται ταχύτατα. 12,5 εκατομμύρια τόνοι θα συλλεγούν. Αυτά τα ηλεκτρικά, ηλεκτρολογικά πρέπει να συλλέγονται και να γίνεται επένδυση σε αυτά. Διότι υπάρχουν σπάνια μέταλλα εκεί και αν μείνουν να έξω επιβαρύνεται και αφαιθούν ελεύθερα επιβαρύνεται το περιβάλλον. Οι συσκευές αυτές θα πρέπει να συλλέγονται και να αξιοποιούνται βάσει συγκεκριμένων μεθόδων. Αλλιώς τα βαρέα μέταλλα ε, εκλείονται στην ατμόσφαιρα ε, αυτό το βλέπουμε και στο φόνης 30% ποσοστό συλλογής μέχρι τώρα έχει επιτευχθεί αλλά πάνω απ' όλα είναι σημαντικό να μην συλλέγονται αδήλωτα ε, αντικείμενα και να ξέρουμε ακριβώς ότι τα συστατικά δεν θα πρέπει να διαχωρίζονται με επικίνδυνο τρόπο. Ευχαριστώ. Η Ευρώπη τα ρίχνει όλα αυτά στους γείτονες παρά τους ε, κανονισμούς και μολύνεται η Αφρική. Είναι πάρα πολλά τα τοξικά που φεύγουν από την Ευρώπη και είναι ανήθικο αυτό και σε οικονομικό και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Οικονομικό γιατί πολλά από τα στοιχεία αυτά έχουν εισαχθεί στην Ευρώπη και έχουμε πληρώσει ακριβά για αυτά και διασπαθίζομαι κάτι που μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί και σε περιβαλλοντικό επίπεδο γιατί οι χώρες δεν μπορούν αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα τοξικά απόβλητα, τα καίνε και με τεράστιες περιοχές όπως και άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά ε, μολύνονται. Οι καινούργιες προτάσεις άργησαν πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, αλλά δεν έχουν αξία εκτός και αν επιβάλλουμε τις διατάξεις σε κάθε κράτος μέλος σταματώντα τώρα τις εξαγωγές. Αυτό το χρωστάμε στον εαυτό μας, αλλά και στους ε, γείτονες που υφίστανται αυτή την ε, κακή χρήση. panie przewodniczący! nowe zasady kładące nacisk na selektywną Κυρίες και κύριοι, οι νέοι κανόνες για την επιλεκτική συλλογή των απορριμμάτων ηλεκτρονικών συσκευών οπωσδήποτε βοηθούν την ανακύκλωση. Τα νέα μέτρα θα εφαρμοστούν προοδευτικά, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό και έτσι τα κράτη θα έχουν χρόνο για να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες. Είναι μεγάλη επιτυχία και το έχουμε πει σε αυτή την αίθουσα το γεγονός ότι υπάρχουν σημεία συλλογής ε, σούπερ μάρκετ ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτό είναι σημαντικό. Ε, εισάγεται με τη νέα ρύθμιση και είμαι πραγματικά ικανοποιημένο από αυτή τη ρύθμιση. Η Πολωνική Προεδρία και το Ευρωκοινοβούλιο συζήτησαν ένα συμβιβασμό. Ισορροπημένο θα έλεγα. Θα προστατεύσουμε την υγεία και η παραγωγή θα επωφεληθούν διότι θα, υπάρχουν, θα υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία. Ο κύριος Γκέρμπραντι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είμαστε στις αρχές του Ιανουαρίου αρχίζουν να παρουσιάζονται αιτήσιες εκθέσεις, γίνονται ε, προγράμματα για την επόμενη χρονιά. Ε, το έτος αυτό θα είναι δύσκολο γιατί υπάρχει ύφεση, ανεργία, πέφτουν οι πωλήσει. Η αυξημένη τιμή των βασικών προϊόντων και άλλων προϊόντων θα επηρεάσει τις εταιρικές χρήσεις. Πολλές ε, έχουν πολύ άσχημα αποτελέσματα, πράγμα που επιβαρύνει την οικονομία επιπροσθέτως. Και αυτό είναι ο πυρήνα τη τωρινή οδηγία, γιατί χάνουμε εκατοντάδε κιλά κοβαλτίου, αργύρου ε, και άλλων πολυτήμων μετάλλων χωρίς να τα ξαναχρησιμοποιούμε. Αυτό λοιπόν πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Ε, το Συμβούλιο ε, δεν βλέπει τι εξοικονόμηση μπορεί να υπάρξει φαίνεται και καθυστερεί. Ευχαριστούμε την Κομισιόν για την εξαιρετική δουλειά για μια συμβιβαστική λύση παράλληλα με την εξαιρετική έκθεση του κυρίου Φλόρεντς. Η ε, συμβιβαστική νομίζω ότι χρειάζεται για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευτυχής και περήφανη που βλέπω το Κοινοβούλιο να καταφέρνει να επιφέρει αλλαγές για μια πιο πράσινη ανάπτυξη και τελικό αποτέλεσμα. Είναι αυτό που πρότεινε η Κομισιόν και ήθελαν και τα κράτη-μέλη. Αυτό ισχύει και για αυτή την έκθεση και για την νομοθεσία που θα συζητήσουμε αργότερα. Χρειάζονται σκληρά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αποτελεσματικά συστήματα ανακύκλωσης. Βεβαίω θέλουμε περισσότερη ανακύκλωση, αλλά τώρα είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Ήδη ακούσαμε για την εξα... τις εξαγωγές ηλεκτρονικών απορριμμάτων και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα γιατί οι χώρες στην Αφρική και αλλού ε, επομίζονται αυτά τα επικίνδυνα απόβλητα. Μιλήσαμε για υπάρχει στις μικρές συσκευέ. Εύκολα μπορεί να συλλεγεί. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αν δεν έχουμε ε, μεθοδή δεν μπορεί να γίνει ανακύκλωση. Ελπίζω ότι θα είναι εδώ καλή η πρόταση της Κομισιόν και βράχει πρόθεσμα. Τρόπο Ποτότσνικ να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο σύντομες απαντήσεις και μία λίγο πιο μακρύ για το ζήτημα αυτό. Για το ζήτημα αυτό δύο μικρές ε, απαντήσεις. Καταρχήν ναι, για τις διαφορές στα κράτη-μέλη. Ναι, είναι τεράστιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται, αλλά είναι σίγουρο 100% ότι οι ευκαιρίες που υπάρχουν είναι επίσης τεράστιες, ιδιαίτερα του χαμηλού επίπεδου οι χώρες. Ε, επίσης για τα συστατικά στοιχεία αυτά ήμουν σαφής. Χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής και θα την έχουν με, στα πλαίσια της σωστής νομοθεσίας. Αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ στα πλαίσια της Κομισιόν. Τέλος ε, για το ιστορικό, γιατί είπα ότι και το περιβάλλον και οι επιχειρήσεις ε, συνεξετάζονται. Αυτή η υπόθεση που προσπαθήσαμε να εξετάσουμε με τον καλύτερο τρόπο με οδικό χάρτη για να έχουμε αποτελεσματικότητα και απόδοση είναι μια κεντρική υπόθεση για το μέλλον της Ευρώπης σήμερα. Πολλές χώρες στην Ευρώπη είναι χρεωμένες στην Ευρώπη. Αν θέλουμε να δώσουμε σωστή απάντηση, δεν θα τη βρούμε αν δεν δώσουμε ενάψματα για την ανάπτυξη. Αν θέλουμε σωστά να απασχοληθούμε με την ανάπτυξη, πρέπει να εστιάσουμε στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αυτά όλα που προτείνουμε, καλύτερη χρήση των πόρων, ε, πιο ευφυής χρήση των πόρων είναι το κεντρικό ερώτημα, το οποίο θα μας βγάλει από τα τωρινά μας προβλήματα. Ελπίζω να γίνει κατανοητό αυτό. Οι τιμές που ανέφερε ο Γκέρμπερ Γιάν ε, αυξάνονται ταχύτατα. Αυτή είναι μια τελείως διαφορετική τάση από εκείνη που είχαμε τον 20ο αιώνα. Οι σύνθετες ε, τιμές των ε, πρώτων υλών έπεφταν τότε συνεχώς με την εξαίρεση του ε, της περίοδου των δύο παγκοσμίων πολέμων και της πετρελαϊκής κρίσης. Ενώ τώρα αντιστράφηκε η κατάσταση ε, και αν λάβετε υπόψη ότι εξαρτάται από εισαγωγές πάρα πολύ η Ευρώπη και αν λάβετε υπόψη ότι στην διάρθρωση του κόστους είναι πολύ περισσότεροι παράγοντες που επηρεάζουν από το εργασιακό μισθολογικό. Βλέπουμε τι γίνεται στις επιχειρήσεις. Ε, εστιάζουν από τις καινοτομίες ε, φεύγουν από την παραγωγικότητα της εργασίας και ε, εστιάζουν στην παραγωγικότητα που απορρέει από τους πόρους. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό είναι ένα κεντρικό συστατικό στοιχείο του συνολικότερου προβλήματος της σημερινής ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα ψηφίσουμε ε, μια πολύ βασική νομοθεσία για τον τομέα αυτό, γιατί έτσι το σωστό κομμάτι της βιομηχανίας που προσανατολίζεται προς το μέλλον, ε, σε αυτούς θα δώσουμε σαφή μηνύματα και προσανατολισμούς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι ο στόχος που ετέθη πολύ υψηλά παρέμεινε αμετάβλητος. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω θερμά ολόκληρο το κοινοβούλιο αλλά ιδιαίτερα τον Καρλ Χάινς ε, Φλόρενς ήταν μεγάλη χαρά να συνεργαστώ μαζί του γιατί η ικανότητά του αλλά και η βαθιά κατανόηση του προβλήματος που έχει μας ε, έδωσε τη δυνατότητα να, κάνουμε, έχουμε αγαστή συνεργασία. Ευχαριστώ. Και εγώ κύριε Επίτροπε και ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον ε, εισηγητή, τον κύριο Καρλ Χέινς Φλόρενς να ολοκληρώσει με τα σχόλιά συζήτηση. Κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι θέσατε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Όλοι διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να αρχίσουμε μια τρίτη βιομηχανική επανάσταση στην Ευρώπη αν καταλάβουμε ότι το θέμα της αηφορίας, της διατηρησιμότητας είναι μια μεγάλη ευκαιρία στη βιομηχανία. Μιλήσατε για πόρους και με φέρνετε σε μια σκέψη που την παραμέλησα. Ξέχασα τους ανθρώπινους σπόρους στο γραφείο μου. Κυρία Αφή, ε, επιτρέψτε μου, γιατί πραγματικά δουλέψατε σκληρότατα, με μεγάλη επιτυχία. Είσαστε κεντρική μορφή σε αυτή τη διαδικασία και σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ κύριε Φλόρεντς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση γύρω από την έκθεση Φλόρεντς ολοκληρώθηκε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Παρακαλώ.